ήθελα να σας ενημερώσω ότι όπως ζήτησε ο κύριος Ντέμες Μέκερ στην προηγούμενη Ολομέλεια, έγραψα στις Ισπανικές Αρχές για να ζητήσω πληροφορίες για την ε, ε, κατάσταση ε, στις φυλακές της Μαδρίτης. Έλαβα τις πληροφορίες που, που ζήτησα. Σύμφωνα με τις αρχές της Μαδρίτης τα πάντα έγιναν ε, βάση νόμου και δεν υπήρχε καμία παραβίαση της ισπανικής νομοθεσίας. Θα στείλω την απάντηση στον κύριο Ντέμες Μάκερ και υπάρχει διαθέσιμη φυσικά η απάντηση και στο γραφείο μου για όσων ε, ενδιαφέρονται.